των Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 134.3, εδάφιο 3 του Κανισμού αποφάσισε το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων του 2010 να αλλάξει και μια ολομέλεια στις 26 Ιανουαρίου σε 9 η ώρα να συγκληθεί στις Βρυξέλλες έχουμε δηλώσεις του Προέδρου όσον αφορά και την Επιτροπή, την εκλογή της νέας Επιτροπής κτλ. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη περνάμε τώρα στη συζήτηση για έξι προτάσεις ψηφίσματος για την περίπτωση της Ουγγάντας νομοθέτημα για την απαγόρευση της